χρονιά να έχουμε πιο αυστηρά, πιο αξιόπιστα και πιο διάφανα τεστ στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Καθυστερήσαμε λίγο κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ τιμητικό όμως ότι αναφερθήκατε σε κάθε ομιλητή. Ίσως λοιπόν για εκπαιδευτικούς ε, λόγους να απαντάτε μόνο σε όσους είναι παρόντες ε, όταν κάνετε δευτερολογία σας για να παραμείνουμε και εντός των πλαισίων του χρόνου. Τέλος πάντων τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Κατόπιν περνάμε σε μια άλλη προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με τις μεταφορές τοξικών αποβλήτων προς αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Δίνω τον λόγο στους ε, ερωτώντες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η κυρία Μπέρντερ για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, αν ξυπνούσε κανείς ε, και έβλεπε πω ο πλούσιο γείτονά μα είχε ρίξει τα σκουπίδια του στην αυλή μα, θα ήμασταν έξαλλοι. Αυτό κάνει όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μέρα. Κάθε χρόνο τόνοι τοξικών αποβλήτων πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανατσόμενε χώρες παραβιάζοντα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Περνάνε από κάτι λιμάνια χωρί ελέγχου. Τρία τέταρτα των ηλεκτρικών αποβλήτων δεν ξέρουμε που καταλήγουν και μόνο το 1 τρίτο διατίθεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο μέσος άνθρωπος πετάει τέσσερις ηλεκτρονικές συσκευέ τον χρόνο. Μιλάμε για 500.000 τόνους, τηλεοράσεις, τηλέφωνα κτλ. Και τα μισά από αυτά δεν ανακυκλώνονται και εξαφανίζονται. Και αυτή είναι η χώρα μου μόνο. Η εξαγωγή αποβλήτων που υπόκεινται σε έλεγχο απαγορεύεται σύμφωνα με την νομοθεσία και όμως κάθε έτος έχουμε παράνομες αποστολές που θεωρούμε πως είναι γύρω στους 22.000 τόνους. Η σχετική οδηγία λέει πως τα εξαγόμενα ηλεκτρονικά είδη πρέπει να λειτουργούν. Όμως αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκές επιθεωρήσεις που σαφώς δεν υπάρχουν. Μιλάμε για πράγματα τα οποία περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο, υδράργυρο ε, και άλλες χημικές και πλαστικές ουσίες που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες όταν καίγονται και η καύση είναι συχνά η φθηνότερη μέθοδος για να ανακτηθούν αυτά τα πολύτιμα υλικά καθώς προσπαθούν άνθρωποι από τα σκουπίδια αυτά να βγάλουν λίγα σέντς. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις σκανδάλου αυτού που πλήττουν τους πιο ευπαθείς. Ως Ευρωπαία ντρέπομαι. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για τις απαντήσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Πώς θα κλείσει αυτό το παραθυράκι στην οδηγία αποστολής αποβλήτων. Έχει η Κομισιόν κανένα σχέδιο για τους τόνους αυτούς αποβλήτων που καταλήγουν στις αφρικανικές χώρες. Και πως πρέπει να αναθεωρηθεί ο κανονισμός είναι απλά ζήτημα επιβολής του. Είναι επίγον το πρόβλημα και πρέπει να δράσουμε τώρα. Αναμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα απόβλητά μας φυσικά δεν εξαφανίζονται διαμαγείας. Δυστυχώς ε, καταλήγουν κάπου που κανείς ε, τελικά δεν τα κατεργάζεται. Και πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν πριν από κάποια χρόνια να στέλνουν με παλιά ferry boat τα αυτοξικά τους απόβλητα στην Ινδία παραδείγματο χάρη. Και βλέπουμε να ξεβράζονται τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα στις ακτές. Και στις αφρικανικές χώρες ε, συλλέγονται κάποια απόβλητα και τα ε, χωρίζουν στα συστατικά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν εφαρμόζει τους ε, πολύ καλούς κανόνες ε, που ορίστηκαν ε, το 12 Ιουλίου του 2006. Και βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού ε, πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά δεν το κάνουν κάποια κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει. Δεν είναι τίποτα τα 70 εκατομμύρια τόνοι, είναι ένα σημαντικό ποσό, μια σημαντική ποσότητα και αυξάνει η ποσότητα αυτή. Και κάτι ε, πρόσθετο, εκτός της προφορικής ερώτησης προς τον Επίτροπο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές, ε, συγκεκριμένοι ε, στοποθεσίες για, το, για τα απόβλητα, για την αποθήκευση των αποβλήτων. Και καλό θα ήταν επίσης να γίνουν και κάποιες προσπάθειες να καταλήγουν τα απόβλητα σε συγκεκριμένους χώρους. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν το πρόβλημα, διότι Αλλιώ δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε καμία πρόοδο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ζέμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, βλέπετε πως οι κανονισμοί δεν ε, αγνοούνται μόνο στις τράπεζες αλλά και στον τομέα των αποβλήτων. Έχουμε τον κανονισμό 2006 που δεν λειτουργεί γιατί διαπιστένουμε πως η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται εκτός της Ένωσης, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου βεβαίως δεν τηρούνται οι σχετικές διατάξεις. Και η λανθασμένη αυτή διάθεση οδηγεί σε προβλήματα υγείας του πληθυσμού που ε, σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί και στο θάνατο αρκετών ανθρώπων. Αλλά βεβαίως και η οικονομία χάνει σημαντικούς πόρους κομμάτι της στρατηγικής 2020 είναι η στρατηγική των πόρων και εδώ πέρα ακριβώς θα πρέπει να δούμε τι πόροι βρίσκονται σε αυτά τα απόβλητα. Γιατί έχουμε σχετικά ερευνητικές προσπάθειες έτσι ώστε στο τέλος του κύκλου ζωής το προϊόν να μπορεί να χρησιμεύσει για την ανάκτηση αυτών των πολιτικών ουσιών. Ο συναδελφός σας, ο κύριος Ποτότσνικ, σε μια ομιλία της 7ης Απριλίου φέτος ανακοίνωσε μετά από μεγάλη κυοφορία εντός της Κομισιόν πως θα εκδώσει μία ανακοίνωση Κομισιόν με στόχο ακριβώς αυτό το πρόβλημα, δηλαδή την εφαρμογή και τις καλύτερες επιθεωρήσεις ε, της ε, οδηγίας ε, για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η υπόθεση λοιπόν. Επίσης ε, αναφέρθηκε ο κύριος Ποτότσνικ σε μια υπηρεσία. Ε, έχουμε πάρα πολλές ε, ήδη υπηρεσίες αποκεντρωμένες. Νομίζω θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες ελέγχου των κρατών μελών. Γιατί διαπιστώνουμε πως το πρόβλημα πρέπει να λυθεί σε αυτό το επίπεδο. Τι άποψη έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζέμπερ. Για τρία λεπτά η κυρία Χάση. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, η οδηγία για τα απόβλητα δεν εφαρμόζεται πολύ σωστά. όπως έχει διαπιστώσει και ένα δίκτυο το οποίο παρακολουθεί τις μεθόδους αυτές από το 2002 και μετά. Υπάρχουν και κάποιες ε, προτάσεις ξεκάθαρες που έχουν γίνει. Βέβαια, η Κομισιόν δεν έχει αντιδράσει με το σωστό τρόπο. Εδώ και 10 χρόνια ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξουν αυστηρότεροι και εντελεχέστεροι έλεγχοι και να υπάρξει σχετική νομοθεσία για ευρωπαϊκού ελέγχου. Το 1999 είχαμε την έκθεση Jackson. Κάποιε ελάχιστε απαιτήσει οι οποίε ε, ορίστηκαν. Επίση είχαμε το 2003 την έκθεση τη μεταρρυθμίσει και το 2008 ένα ψήφισμα για τους ε, ελέγχους και τις ελάχιστες απαιτήσει που πρέπει να πληρούν. Αγνοήθηκαν όλοι αυτοί, όλες αυτές οι εκθέσεις από την Κομισιόν. Ουσιαστικά το 2006 υπήρξε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο με την τρανσφίγκουρα. Στην ακτή του Λεφαντοστού κατέληξαν ε, μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και τότε ο Επίτροπος ε, Δήμας είχε προτείνει ε, είχε πει ότι θα βρει τρόπους για να διορθωθεί η κατάσταση και υπήρχε ο κανονισμός για τις εξαγωγές και την υλοποίησή τους για τα κράτη-μέλη. Δεν έγινε όμως κάτι συγκεκριμένο. Πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες μελέτες που έκανε ε, διαπίστωσε ότι πρέπει να συγκροτηθεί ένας φορέας που θα αναλάβει την, εκτέλεση, την εποπτεία της εκτέλεσης του των ρυθμίσεων για τη μεταφορά αποβλήτων. Παραδείγματο χάρη έλεγχη στα κράτη-μέλη, συντονισμό των ελέγχων, αλλά δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη πρόταση παρόλα αυτά. Πέρυσι, μια μελέτη της Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη εναλλακτική λύση θα ήταν να υπάρξει μια νομική πράξη που θα θέτει τα κριτήρια για τους έλεγχους. Πάλι δεν έγινε τίποτα συγκεκριμένο. Μας λέει η Κομισιόν όμω ότι ε, ο Επίτροπος συγκεκριμένα μας λέει ότι είναι προτεραιότητά του εφαρμογή της παραγωγικής Σε Ερωτώ λοιπόν. Πότε θα αναλάβει ε, δράση η Επιτροπή πάβοντα τι μελέτες πια. Πότε θα έχουμε συγκεκριμένες νομοθετικέ προτάσεις και όχι ανακοινώσει και μελέτε. Όπως είπε και ο κύριος ε, Ζέιμπερ, αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πόρων στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κυρία Χάση. Τελευταία από τους ερωτώντες η κυρία Βίλση, για δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παράνομη μεταφορά αποβλήτων κινδυνεύει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και απειλεί και το περιβάλλον. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται συνεχώς τα τοξικά απόβλητα λόγω του υψηλού κόστους ε, και άρα είναι μεγάλος ο πειρασμός να τα στείλουμε όλα αυτά σε χώρες με χαμηλότερο κόστος διάθεσης. Χαίρομαι για το ότι το πρόβλημα αυτό το είδαμε και το αναγνωρίσαμε διακομματικά και ελπίζω το Κοινοβούλιο να δράσει εδώ από κοινού. Τα κενά στην ομοθεσία που επιτρέπουν τη δηλητηριώδη αυτή εξαγωγή πρέπει να κλείσουν. Υπάρχουν κανονισμός, πρέπει να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί. Χρειαζόμαστε μια νομοθετική πρόταση για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που είχε ζητήσει ήδη το 2008 το Κοινοβούλιο έτσι ώστε τα πλοία να ελέγχονται στα λιμάνια από τις επιτόπου αρχές. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα τα πλοία όταν υπάρχει αιτιολογημένη υποψία να μπορούν να τα σταματάνε στα λιμάνια. Εμείς προτείνουμε να μπει αυτό σε ένα κοινό ψήφισμα όλων των ομάδων και η διάθεση των αποβλήτων στην Ένωση πρέπει να ελεγχθεί καλύτερα. Στην ακτή της Καλαβρίας λίγα μίλια από το λιμάνι Σεντράρο είναι βυθισμένο ένα πλοίο το οποίο μετέφερε δηλητήρια και άλλα υποθέτουμε πως είναι βυθισμένα στις τυρινικές ακτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια και αξιόπιστη κρατική έλεγχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βίλς. Ξονόματος της Κομισιόν ο Επίτροπος ο κύριος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ποτότσνικ είναι στη Νέα Υόρκη για την υπογραφή μιας σημαντικής σε για τη βιοπικιλότητα και εκφράζει τη λύπη του ε, Διεμού που δεν μπορεί να παρίσταται εδώ σήμερα. Ελπίζω να μπορέσω να τον αναπληρώσω, διότι είναι και ένα θέμα που πάντοτε με ενδιαφέρε. Ήμουν και υπουργό περιβάλλοντος στη χώρα κατά το παρελθόν και όταν πρώτο ανέλαβα τα καθήκοντα του Επιτρόπου πριν από 10 χρόνια, είχα και εγώ βοηθήσει μαζί με το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει η αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματο. Ο κανονισμό λοιπόν για τη μεταφορά ε, αποβλήτων απαγορεύει τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρε καθώ και τι εξαγωγέ ε, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών ΑΕΛΕ, των χωρών ΕΖΕΣ δηλαδή. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί η απαγόρευση, αλλά ποικίλουν οι προσπάθειες αυτές από το ένα κράτος στο άλλο. Πολλές φορές ε, οι φορείς υποφελούνται ε, της έλλειψης επαρκών ελέγχων για να παρακάψουν ε, τους ελέγχους και να μεταφέρουν μέσω άλλων κρατών μελών τα απόβητα σε άλλα κράτη τα οποία λοιπόν δεν έχουν τόσο αυστηρούς ελέγχους και με ψευδείς δηλώσεις πηγαίνουν αυτά τα απόβλητα ως μεταχειρισμένα προϊόντα ή κάτι άλλο, πηγαίνουν στις ε, τρίτες χώρες. Και βέβαια υπάρχει και ένα πολύ χαμηλό κόστος επεξεργασίας στις τρίτες χώρες. Αυτός είναι ένας οικονομικός παράγοντας που ευνοεί παροτρύνει πολλούς να προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες μεταφορές. Και υπάρχει βέβαια και μια σοβαρή κατάσταση των κρατών που λαμβάνουν αυτά τα απόβλητα μέσω αυτών των παράνομων μεταφορών που οφείλονται στην ε, ρήπανση του αέρα, των ε, εδαφών, ε, του νερού. Όπως είπατε κυρία Βίλσε και όπως είπε και η κυρία Μπέρντερ και η κυρία Ρόσμπαχ, ουσιαστικά απειλούν την υγεία των ανθρώπων, την υγεία των παιδιών. Αυτό είναι σκανδαλώδε. την υγεία των εργαζομένων. Μεγάλο μέρο του πληθυσμού πλήττεται από την πρακτική αυτή. Επίση σε κάποια στόξικέ ουσίε που έχουν αυτά τα προϊόντα αποτελούν ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Και φυσικά δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία για την αντιμετώπιση, για την επεξεργασία αυτών των αποβλήτων στι ε, περισσότερε από τι χώρε υποδοχή. Δεν μεταφορά αποβλήτων ε, στι ε, τρίτε χώρε χώρες επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Διότι από οικονομικής πλευράς οι επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται την νομοθεσία τελικά θίγονται και αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Η ανακύκλωση ή η διαχειριση των αποβλήτων που πρέπει να τηρεί τις αυστηρές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας 95 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο κύκλος εργασιών 1,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 1% του ΑΕΠΑ. Αυτός ο τομέας λοιπόν της διαχείρισης των αποβλητών της ανακύκλωσης που εργάζεται σωστά και αυτός πέφτει θύμα ανταγωνιστικού μειονεκτήματος λόγω αυτής της παράνομης μεταφοράς. Εάν εφαρμοστεί όμως σωστά η νομοθεσία, νομίζω ότι θα εμφανιστεί ο τομέας να επενδύσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Διότι αν υπάρξει ανακύκλωση κακών προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται και πρώτες ύλες. Και δεν καλύπτονται οι ανάγκες σε πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Ενώ αν ισχύσουν οι κανόνες θα μπορεί να γίνει μια πιο χρηστή διαχείριση των πόρων. Θα πρέπει λοιπόν με βάση τη διάγνωση αυτή της κατάστασης να προβούμε σε βελτιώσεις. Γι' αυτό και στην Κομισιόν ε, προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσο πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα σε επίπεδο ένωσης και ενδεχομένως να δούμε ποιε απαιτήσει και ποια συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίσουμε για τους ελέγχους που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά αποβλήτων. Ολοκληρώνεται μία μελέτη επιπτώσεων αυτόν τον ε, καιρό για να λυθεί το ζήτημα το οποίο ανέφερα. Ε, τα εθνικά προγράμματα ελέγχων, αξιολόγηση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι υποχρεωτική και επίσης ε, η σωστή εκπαίδευση, πιο στοχευμένη εκπαίδευση των επιθεωρητών και να υπάρξει και αναστροφή του βάρους απόδειξης για αυτούς που κάνουν ψευδείς δηλώσεις των αποβλήτων λέγοντας ότι πρόκειται για μεταχειρισμένα προϊόντα. Τώρα, ολοκληρώνοντας να απαντήσω σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να παρακαμφθεί ο κανονισμός της μεταφράσης τοξικών αποβλήτων αν ε, υποστηριχθεί ότι είναι μεταχειρισμένα τα προϊόντα και όχι απόβλητα. Το πρόβλημα είναι ότι τελικά δεν εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη-μέλη η απέτηση που αφορά του ελέγχου. και έτσι θα μπορούσε να διορθωθεί το πρόβλημα. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί με πιο αναλυτικούς κανόνες για τους εθνικούς ελέγχους. Για τα νομοθετικά τώρα μέτρα, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται με κατάλληλη εκπαίδευση των αρμοδίων για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων. Τώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη δεσμευτικέ νομικά ε, κατευθύνσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν, τον έλεγχο της εφαρμογής ε, του κανονισμού για τη μεταφορά των απολύτων μέσω των τελωνίων συγκεκριμένα και έτσι θα καταπολεμηθούν παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν θα αρκέσουν οι απλές κατευθυντήριες γραμμές, θα χρειαστούν και δεσμευτικοί κανόνες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Τώρα, συνολικά και έρχομαι στο τρίτο μου σημείο, η παραγωγή αποβλήτων έχει αυξηθεί ή σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η διαχείριση των αποβλήτων βελτιώνεται στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Η ανακύκλωση τα πέντε τελευταία χρόνια αυξήθηκε. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο σήμερα ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων για τα απόβλητα. Έχει επίγνωση κομισιών των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, ανθρώπινων επιπτώσεων, επιπτώσεων για την υγεία, τη δημόσια υγεία, που μπορεί να έχουν η παράνομη μεταφορά τοξικών αποβλήτων. Και ξέρουμε ότι πολλοί εκτέθηκαν σε ε, σε αυτά τα απόφυτα τα οποία αναφέρατε, τα οποία ε, ξεβράστηκαν σε ακτές ακτές του ελεφαντοστού και έχουν γίνει πολλές μελέτες για το θέμα. Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας τα σχετικά αποτελέσματα τώρα. Από τη στιγμή που εντοπίζεται παρανομή μεταφορά ενό αποβλήτου, προβλέπονται διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να, παρα... να αναπευθούν στη χώρα προέλευση βάσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτά τα απόβλητα και βάσει του διεθνού δικαίου. Αν τώρα οι αρμόδιες, οι υπεύθυνε εταιρείε ε, δεν μπορούν να βρεθούν, τότε θα πρέπει να υπάρξει τιμολόγιο για τον επαναπατρισμό αυτών των αποβλήτων και ίσως κάποια κράτη-μέλη ε, χρειαστεί να πληρώσουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, όπως στην περίπτωση αυτή του Προμπόκο, αλλά στην περίπτωση αυτή δηλαδή της ακτής ελεφαντοστού που σας προανέφερα. 152 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έξοδα για τον καθαρισμό και 33 εκατομμύρια ήταν η αποζημίωση για τους κατοίκους των περιοχών που ε, πλήγησαν. Θέλω να πω επίσης την καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ποτότσιν έχει δεσμευθεί να κάνει αυτή την ανακοίνωση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και μάλιστα την εκπονή. Αυτό ήθελα να σας ε, πω αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις ομάδες. Μόνο μία παρέμβαση έχουμε από τον κύριο, την κυρία Βέστελουντ για τρία λεπτά. Eh, Ευχαριστώ. Ξέρετε πως ε, είναι λυπηρό το ότι πρέπει να γίνει άλλη μία συζήτηση για την απόρριψη των τοξικών αποβλήτων και πάρα πολύ είναι οργισμένοι. Χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία διαταράσσουν το περιβάλλον και έχουμε μετά απόβλητα που βλάπτουν την υγεία των παιδιών, τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ότι μπορεί δηλαδή να συνεχίζεται. Υπάρχει νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται, άρα η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει αλλαγές. Βεβαίως, καλό θα είναι να μην ε, χρησιμοποιούσαμε καν τέτοιες επικίνδυνες χημικές ουσίες και το προσπαθήσαμε με το ΡΙΤΣ. Εξαγωγή λοιπόν δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται και άρα έχουμε και ισχυρή νομοθεσία συλλογή των αποβλήτων. Υπάρχουν όμως λόγοι για τους οποίους η Κομισιόν θα πρέπει να δει τι κάνουν τα κράτη με τη σχετική οδηγία. Η Κομισιόν είπε πως χρειάζεται διευκρίνηση και απλοποίηση των διατάξεων όσον αφορά την διάθεση αποβλήτων έτσι ώστε αστυνομία και συνοριοφύλακες να βλέπουν αν υπάρχουν περιβαλλοντικά εγκλήματα θα πρέπει λοιπόν να είναι αυτό μία πρώτη προτεραιότητα. Δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους τα κράτη-μέλη περί ελέγχου. Και είναι σαφές αυτό. Πρέπει να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη και αναμένουμε να το κάνει αυτό η Κομισιόν. Δηλαδή. Και Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπαρνιέ είναι προς σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε πως θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ευχαριστούμε κυρία Βέστλουντ. Περνάμε στην οφθαλμοθυρική διαδικασία, κυρία Ρόιτοβα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γιατί φαίνεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ορολογιακή βόμβα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου εξάγουμε τοξικά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα σε τεράστιες ποσότητες. Καλωσορίζω, Επίτροπε, την δήλωσή σας όταν λέτε ότι η Κομισιόν θέλει να καλύψει τα κενά τα οποία υπάρχουν στην νομοθεσία και αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχω όμως την εντύπωση ότι, υπάρχει, ότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση στα κράτη-μέλη. Δεν θέλουν να επιβάλλουν νομοθεσία, δεν θέλουν να επιβάλλουν τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίαση των ισχύου, της ισχύουσας νομοθεσίας Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εκπονήσουμε και μια κοινή στρατηγική με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, τις χώρες ΑΚΕ, ε, για να υπάρξει ένα σύστημα ασφαλούς διαχείρισης ε, των τοξικών αποβλήτων και κυρίως να προωθήσουμε την ανακύκλωση των αποβλήτων. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αυστηρή. Στην πράξη όμως υπάρχουν παραθυράκια και η μαφία τα εκμεταλλεύεται. Και η μεταφορά τοξικών αποβλήτων είναι καλή μπίζνα. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι το υψηλό κόστος ε, ανακύκλωσης. Ο άλλος λόγος ε, είναι πως είναι πολύ γραφειοκρατική η διαδικασία. Αφενός, άρα θα πρέπει να μειώσουμε το κόστος της νόμιμης ανακύκλωσης και το διοικητικό βάρος και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται νόμιμα. Από την άλλη να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι και κυρώσεις κατά της μαφίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σέγγεντη. Για ένα λεπτό κύριος Νικολάσικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 12 ε, Κοιτάξτε, είναι σχεδόν μεσάνυχτα και συζητάμε ένα πολύ σοβαρό θέμα Μιλάμε για την μεταφορά τοξικών αποβλήτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ένα σκανδαλώδες 21ο αιώνα οι ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν πράγματα τα οποία κάναμε, που βλέπαμε σε ταινίες με την Έριν Μπρόκοβιτς, την, την Τζούλια Ρόμπερτς να δίνει τη μάχη αυτή. Εμείς θεωρούσαμε μονάχα στην Καλιφόρνια γίνονται όλα αυτά τα θέματα με τοξικά απόβλητα και με θανάτους κτλ. Είναι λυπηρό οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξάγουν τοξικά απόβλητα σε αφρικανικές χώρες. Οι χώρες αυτές δεν μπορούν να προστατευτούν. Έχουμε επικίνδυνες ε, ε, χημικές ουσίες, ε, υδράργυρος, μόλυβδος, ουσίες που είναι ιδιαίτερως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Χαίρομαι που ο Επίτροπος μας προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και ελπίζω ότι αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μακίνες. Thank you, Mr. President. Um, there's a problem... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, στη, στο κατόβλη του σπιτιού μας πετάμε τα ε, σκουπίδια αυτά και τα απόβλητα. Ό,τι και να κάνουμε ε, σίγουρα είναι ε, πάρα πολύ καταδικαστέα αυτά τα οποία γίνονται με την ε, ε, απόρριψη αποφύγων σε τρίτε χώρε. Ε, είπατε για νέα νομοθεσία, αλλά νομίζω ότι το, και φοβάμαι ότι απλά θα δημιουργήσουμε ένα στρώμα παραπάνω, αλλά δεν θα δούμε την, την εφαρμογή και την επιβολή αυτής της νομοθεσίας. Σας παρακαλώ λοιπόν να αντιμετωπίσετε και αυτό το θέμα τη επιβολή τη νομοθεσίας. Νομίζω ότι σε πολλέ περιοχέ δεν υπάρχουν αρκετό προσωπικό για να ελέγξει τη μεταφορά αποβλήτων και συγκεκριμένα τοξικών στην προκειμένη περίπτωση και οι συνέπειες για την υγεία, για την ευημερία και αυτών που χειρίζονται τα απόβλητα με πολύ κατάλληλο τρόπο είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα θέμα ηθικής δεοντολογίας και ίσως αν το γνώριζαν οι συμπολίτε μας, δεν νομίζω να το γνωρίζουν, αλλά αν το γνώριζαν ίσως να το ξανασκέφτονταν για τις μεθόδους ε, αγοράς και διάθεσης. Σας ευχαριστώ κυρία Μακίνες ο κύριος Επίτροπος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Μικρόφωνο. θα ακολουθήσω τη σύστασή να είμαι σύντομος. Η κυρία Μαγκίνες είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησε για την ηθική με όλες αυτές τις ανησυχίες για την δημόσια υγεία, για την βιοπικιλότητα, για την οικονομία γενικότερα. Γι' αυτό και στην κυρία Βέστρουν και στην κυρία Ρόιτεβε και σε στους άλλους ομιλητές ότι η Επιτροπή είναι ε, αποφασισμένη να δράσει και με την υποστήριξή σας η Κομισιόν θα προτείνει μια ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κυρίως για να βελτιώσουμε τους ελέγχους ε, ε, για την μεταφορά των αποβλήτων και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα περιορίσουμε τις παράνομες μεταφορές. Όλες οι λύσεις εξετάσσονται. Να πω στον κύριο Ποτόσνικ ότι ε, υπάρχουν κάποιες εβδομάδες που θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να, και μιλάω εξ ονόματος του κ. Ποτόσνικ, ότι ε, χρειαζόμαστε κάποιες ομάδες για να προετοιμάσουμε την νομοθεσία. Ε, τέλος πάντων, θα υποβάλουμε προτάσεις στο, άμεσο μέλλον για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτές τις παράνομες μεταφορές οξυγόνων προβλήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ όσους έμειναν μέχρι τα μεσάνυχτα. Α, υπάρχει αυτή κάπως